Thank Σας ευχαριστώ όλους. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, πάνω στην ώρα, μετά την καθυστέρηση φαίνεται ότι είμαστε στην ώρα μας και περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ετήσια έκθεση για το 18-19. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κλέρ Ντέιλι από τη Γκουε. Θα δούμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης. Έχετε το λόγο και μετά θα γίνει συζήτηση εάν υπάρχουν ε, μέλη που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρουσιάζω το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μέγαν Κέλλιεν και τη, ένα μέλος ε, της ομάδας Μεξικού, ένα άλλο μέλος, ε, δυστυχώς πολλές φορές δεν τους αποδίδουμε τα εύσημα που αξίζουν. Γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την εργασία τους. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, ήταν ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα χρόνια μετά όμως θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχει εφαρμοστεί και τι πρέπει να αλλάξουμε έτσι ε, ώστε η χάρτα, ο χάρτης να είναι μια απτή πραγματικότητα. Και γι' αυτό καταρτίστηκε αυτή η έκθεση στα πλαίσια της ε, εργασίας της Επιτροπής, η Επιτροπή ακριβώς προβαίνει σε μία ε, αναθεώρευση μετά από την ε, πρώτη δεκαετία λειτουργίας αυτού του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς. Είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση με τους σκιώδεις, όπου θελήσαμε να έχουμε μία πιο συνεκτική έθεση. Ξέρουμε ότι αυτά που επιθυμούμε και αυτά που επιτυγχάνουμε δεν ε, ταυτίζονται, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν έχουν αναφερθεί τα πάντα διεξόδικα. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε τα ζητήματα που δεν έχουν αναφερθεί, αλλά θεωρούμε ότι η Επιτροπή μας έχει αναλάβει έργο και σε άλλους τομείς το 2020 ως προς το κράτος δικαίου για παράδειγμα, οπότε δεν υπήρχε λόγος για επικάλυψη. Εμείς θελήσαμε να εστιάσουμε την προσοχή σε τομείς όπου δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, απειλούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το γράμμα του χάρτη δεν έχει εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς. Ε, ως προς το ρατσισμό, ξενοφοβία, ισλαμοφοβία, βία κατά των προσφύγων και των ασύλου, κατά των μεταναστών και κατά του τύπου δεν χρειάζεται να είναι κανείς, ε, να είναι για να αναγνωρίσει το εύρος των προβλημάτων. Θα πρέπει να δούμε όμως γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, ίση μεταχείριση, δικαιώματα ε, και καθήκοντα των μεταναστών και των προσφύγων μεταξύ άλλων. Μερικά ζητήματα ε, υπερεκτιμώνται ή τονίζονται περισσότερο σε αυτή την έκθεση. Ξέρω ότι άλλες ομάδες δεν θα μπορούσαν να συνδράμουν πάντα σε όλους τους τομείς, αλλά ήθελα να σταθώ στα ευρύτερα ζητήματα που μας απασχολούν ως προς τις ελευθερίες και την ίση μεταχείριση τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα διονγκούνται. Και ήθελα και ε, οι άλλοι συνάδελφοι να ασχοληθούν με όλους τους τομείς σε σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι ύψης της σημασίας, ε, πολλές φορές είναι θέματα που βρίσκονται εκτός εκτός εθνικής, ε, εθνικού πλαισίου. Θα πρέπει να δούμε όμως, ε, θα πρέπει να δούμε την ουσία. Αν δεν έχει κανείς ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του ή δεν έχει να φάει, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ζητήματα ουσίας που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσουν. Και ξέρουμε ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες ως προς το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, το αντιμετωπίσαμε το ζήτημα λίγο διαφορετικά, δηλαδή μιλάμε για αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, ένα ευρύτερο φάσμα. Αλλά αν δείτε την ε, ε, διάκριση κατά τον Ρωμά, στην οποία πάντα αναφερόμαστε, τι σημαίνει αυτό. Ε, λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, το τονίσουμε ότι δηλαδή οι γυναίκες Ρωμά ε, έχουν διαφορετική μεταχείριση και χώρους στα νοσοκομεία. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τουαλέτες, τα ίδια δωμάτια και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και τον διαχωρισμό αυτό, τον εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρωμά ε, μια, ένας άλλος τομέας ασχολείται με τις ελευθερίες, το ε, δικαίωμα τα, τις ελευθερίες του τύπου, το δικαίωμα του ε, συνέρχεσθε. Γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση ως προς το μεταναστευτικό και τους ετούντες άσυλο και θα έπρεπε να συμπαραταχθούμε και ε, με αυτό το τομέα ως προς τα δικαιώματα των μεταναστών και των ετούντων άσυλο και των προσφύγων. Πρόκειται για μια συνοπτική εικόνα έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να βάλουν το δικό τους ε, input και εμείς ε, θα προβάλλουμε τροπολογίες και ελπίζω να το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, πιστεύω ότι θα έχουμε να κάνουμε με ένα συλλογικό εγχείρημα, να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κατιεράρχηση θέματα, Διαφορετικά δεν επιτυγχάνουμε τίποτα και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ορισμένους τομείς γιατί βρισκόμαστε στο δέκατο έτος εφαρμογής και ευχαριστώ πολύ και τους, και τους υπαλλήλους που βοήθησαν στη, στη σύνταξη αυτή της έκτασης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέλη. Ας τα συζητήσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις και μετά όποιος άλλος βουλευτής θέλει να πάρει το λόγο. Έχουμε λοιπόν καταρχήν τον ε, Κάρλο Ρέχσλερ ως πρώτο ομιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια αλλά να την εξηγήσω και για την επεξηγηματική έκθεση που προσπάθησε να διευκρινίσει κάποιες από τις θέσεις όταν συζητάμε την κατάσταση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καμιά φορά είναι εύκολο να υπονομεύσουμε κάποια τμήματα, να τα μειώσουμε, να ε, ε, φωτίσουμε υπερβολικά κάποια άλλα. Ε, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εστιάσουμε στα σημαντικά και πιστεύουμε το ότι μια τέτοιου είδους επίσημη έκθεση θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, αλλά παράλληλα να προσπαθήσει να ακολουθήσει και μια ολιστική προσέγγιση για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ευρύ και περιγράφει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάποια συγκεκριμένα θέματα πιστεύουμε πως θα πρέπει να αναφέρονται, το έκανε η συγγήτρια, εκεί που επηρεάζονται, όπως η κατάσταση των προσφύγων, όπως επίσης των Ρωμά, αλλά και των ειρηνικών διαδηλωτών. αλλά με το να αποκλείουμε ε, κάποιες ολόκληρες περιοχές όπου έχουμε αρνητικές επιπτώσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα ή δυνητικά θα μπορούσαν αυτά να επηρεαστούν αρνητικά, στέλνουμε ε, ε, το λάθος μήνυμα στις ευάλωτες ομάδες. Γι' αυτό εμείς ως προτεραιότητες τονίσαμε αρκετούς τομείς στους οποίους θα θέλαμε να, οποίους θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Καταρχήν, ευάλωτες ομάδες δικαίωμα και ελευθερίες οι οποίες ε, πλήττονται ε, λόγω των διεθνών και σύγχρονων προκλήσεων. Στα τροπολογία που θα επιβάλλουμε λοιπόν θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ευάλωτες ομάδες για την ανθρωπιστική κατάσταση και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη για διατύπωση η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες για την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των μεταναστών. Αλλά εδώ θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και τη μάχη κατά των διακινητών ε, του τράφικινγκ Και να σας πω το εξή. Έχουμε τεχνολογική και ψηφιακή πρόοδο η οποία βοηθά, αλλά δεν έχουμε την απαραίτητη ρυθμιστική δράση για τα θέματα, με αποτέλεσμα τα θεμελιώδη δικαιώματα να επηρεάζονται με αρκετούς τρόπους. Κυρίως όταν παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα ή ο ιδιωτικό χώρος των πολιτών μας. Τέλος, η σχετική υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρεται στον αντισημιτισμό σε μία από τις μεγάλες προκλήσεις. Οι πολίτες μας στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουν σήμερα και εκεί προτείναμε να το καλύψουμε στα πλαίσια της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεπιθήσεων, της ελευθερίας της έκφρασης, συγκέντρωσης και ε, σκέψης. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτό να καλύπτεται απόλυτα στο πρώτο σχέδιο έκθεσης, αλλά καλωσορίζω πραγματικά γιατί καταλαβαίνω πως έχει δεσμευθεί η εισηγήτρια να το καλύψει αργότερα. Αυτές θα είναι περίπου οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Με χαρά περιμένω να συνεργαστώ μαζί σας και από εμάς να σας πω πως η έκθεση αυτή θα πρέπει να είναι λίγο πιο ισορροπημένη, λίγο πιο ολιστική και συνολική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρέσλερ, εισηγητή του ΕΛΚΑ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ίνσνερ από τους σοσιαλιστές. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τη γραμματεία γιατί εξαιρετικά πετυχημένη δουλειά που έχουν κάνει, όπως επίσης τους ε, σκιώδες για τη συνεργασία. Δεν νομίζω πως ε, χρειάζεται να το πω, παρόλα αυτά θα το επαναλάβω. Η δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου δεν είναι δεδομένα τουλάχιστον αυτούς τους ε, καιρούς που βλέπουμε να κινδυλεύουν όλα σε κάποιες χώρες. Κάτι το οποίο μεταδίδεται δυστυχώς και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές και διαφορετικά δεν θα το δεχτούμε τώρα. Η εισηγήτρια μίλησε πολύ σωστά. Είναι σύντομη η εισήγηση, είναι, ε, συγκεντρώνεται και εστιάζει στα βασικά θέματα και είναι και προσιτή. Μπορεί να την διαβάσει κανείς εύκολα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λόγια της ε, στην καθημερινή μας δουλειά. Όπως είπε και ο συνάδελφος, στην έκθεση έχουμε συγκεκριμένα σημεία που είναι εξαιρετικά, αλλά έχουμε και κάποια άλλη που για μένα υπάρχει χώρος βελτίωσης. Όπως φαντάζεστε, εμείς οι σοσιαλδημοκράτες θεωρούμε πως τα κοινωνικά δικαιώματα είναι απαραίτητα και θα πρέπει να συνδυάζονται με τα θεμελιώδη βασικά δικαιώματα. Έχουμε ε, κάποια βελτίωση σε αυτό αλλά η συγγήτρια εστιάζει στα κοινωνικά δικαιώματα και λιγότερο σε άλλα δικαιώματα, τα οποία επίσης, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπογραμμιστούν περισσότερο. Επαναλαμβάνω, λόγω των καιρών στους οποίους ζούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο νομισματική ένωση, είναι και κοινωνική για τους ανθρώπους και όχι μόνο για τα κεφάλαια. Πολύ σωστά το λέει η έκθεση. Αλλά είναι ένωση που βασίζεται σε κοινέ αρχές. Το λέει το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Επίσης, τέτοιου είδους εκθέσεις πολλές φορές αποτελούν απλώς μία, ένα κατάλογο χωρών που δεν σέβονται τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα, άλλα πιο σοβαρά, άλλες παραβιάσεις λιγότερο. Οπότε θέλουμε και άλλες πληροφορίες. Ποιος ε, κατά και με ποιο τρόπο. Αλλά για να μην έχουμε μία απλή παράθεση, θα πρέπει να εξηγούμε γιατί συγκεκριμένε χώρε αναφέρονται και άλλε όχι. Στο τρέχον σχέδιο, εγώ δεν βρίσκω να υπάρχει αυτό. Και μία τέτοια έκθεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με κομματικούς ε, σκοπούς. Και το λέω αυτό γιατί ως νέα ευρωβουλευτής έχω βαρεθεί από τις συζητήσεις που γίνανε πέρσι και κάποιες ομάδες δεν θέλουν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα των όσων συμβαίνουν σε κάποιες χώρες. Δεν μιλάμε μόνο για μεμονωμένες υποθέσεις. Δυστυχώς στην Ευρώπη δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις η παραβίαση σε κάποιες περιπτώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί συστηματική παραβίαση ε, κάποιων θεσμών ε, και οι θεσμοί αυτοί που ε, καταλύονται είναι οι θεσμοί ακριβώς που μας προστατεύουν εμάς και τα δικά μας δικαιώματα. Η έκθεση αναφέρεται πολύ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο πολιτικό αλλά και στις μη πολιτικές του ε, δομές. Εδώ ίσως θα έπρεπε να αναφερθούμε και στα δικά μας, ε, στις δικές μας υπηρεσίες σχετικές με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αν δεν μιλάμε για τους δικούς μας θεσμούς εμείς, ποιος θα το κάνει στη θέση μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτά να τα συνδέσουμε ε, με τη δουλειά που έχει κάνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Βιέννη. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθούμε σε διάφορες φοβίες. Ισλαμοφοβία, αφρικανοφοβία, τρομοκρατικές επιθέσεις πέρσι ε, που προέρχονται από τέτοιου είδους φοβίες, η χθεσινοί όπου ε, επιτίθονται κατά ομάδων λόγω ε, καταγωγής ή θρησκευτικών πεπιθήσεων. Έχω κι άλλα να πω. Οι τροπολογίες μου θα βασίζονται και στα στοιχεία τα οποία ανέφερα και σε κάποια άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, από την ομάδα Renew, η κυρία Παγάσα Ορτοντούα είναι σκιώδη, αλλά δεν ξέρω ποιο θα την αντικαταστήσει. Η κυρία Νετφέλτ, μάλιστα από το Ρινιού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω αυτά που μου άφησε η συνάδελφος και θα προσθέσω δύο-τρία πραγματάκια δικά μου. Η κυρία Παγάσα Ορτουντούα λέει κατά τη γνώμη της η έκθεση δεν ανακλά ικανοποιητικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση ως προς τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι μια βάση για ε, συνεργασία και για εργασία, αλλά χρειάζεται κάποιε αποχρώσεις που θα φέρουν άλλες πολιτικές ομάδες. Ε, τονίζονται κάποια σημεία που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ισότητα, ελευθερία στη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτά χωρί καμιά αμφιβολία είναι σημαντικά και συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κρίσιμα σημεία που είναι εκτό τη έκθεση, όπω οι παραβιάσει των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ή ε, τα δικαιώματα ε, που θίγονται από την παραπληροφόρηση ή ε, την ψηφιακή εποχή. Ρατσισμός, ξενοφοβία, διακρίσεις, ρητορία μίσους παραγνωρίζονται και είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι θεωρούνται πλέον κανονικά, φυσιολογικά όλα αυτά. Στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να τονιστούν περισσότερα. Αντίθετα, είναι ιδεολογικά φορτισμένη η έκθεση και αυτό το βλέπουμε σε ιδεολογικές σκέψεις. Ε, τέτοιου είδου εκθέσει θα πρέπει να βάζουν τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω θεσμικό όργανο, να στέλνουμε σημαντικά ε, μηνύματα στα άλλα θεσμικά όργανα, στα κράτη-μέλη και στου πολίτε. Ε, θα κάνω τροπολογίες, λέει η κυρία Παγάσα Ορτοντόα, για να συμπληρώσουμε την έκθεση και να διευκρινίσουμε κάποιες από τις προτάσεις. Αυτά λέει η δική μας σκιώδης συγγήτρια. Και τώρα θέλω να προσθέσω μερικά σύντομα σχόλια ως Init Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάνουμε πολλή ενέργεια ε, και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί ένα ευχολόγιο θα είναι η έκθεση, όπως συνήθω είναι. Δεν πειράζει. Ο καθένας έχει τις δικές του προτεραιότητες. Αυτό εμπλουτίζει την έκθεση. Ε, το σχέδιο έκθεσης πραγματικά ε, περιορίζεται σε κάποια μόνο θέματα. Είναι γεγονός αυτό. πώ να το πω. Είναι πολιτικά φορτισμένο, ιδεολογικά ε, μεροληπτικό. Τι να κάνουμε, πολιτικές ομάδες έχουμε, πολιτικοί είμαστε. Σε εμά εναπόκειται να κάνουμε τροπολογίε ως Επιτροπή και προσβλέπω στην ευελιξία τη εισηγήτριας για να διαπραγματευτούμε καλέ συμβαστικέ τροπολογίες. Τώρα θα πρέπει να κατονομάζουμε και να διαπομπεύουμε χώρες, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας ευρύ μηχανισμός για τη δημοκρατία, κράτο δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει κάτι με πιο στενό πεδίο. Εμείς ζητήσαμε συστάσεις ανά χώρα. Τώρα, όσο είναι δίκαιο, γιατί να μην τους κατονομάζουμε, δεν κατάλαβα. Αφού υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά του. Και τέλος, να επαναλάβω και κάτι που είπαν προλαλήσαντες, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που έχουμε στα κράτη-μέλη που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Όπως η ΛΟΑΤΚΙ, η ομοφοβία, ελευθερία του λόγου, ε, παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας και ένα σωρό άλλα θέματα που συνδέονται σίγουρα και με την ε, αύξηση του ακροδεξιού εξτρεμισμού, όπως ακούσαμε και χτες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εισηγήτρια. you, Ευχαριστώ κύριε Νιτβέλτ. Και τώρα η πράσινη. Η κυρία Διάννα Ρίβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία, για την προθυμία της και την καλή εστίαση που επέλεξε. Τα τελευταία δύο χρόνια, στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη έκθεση, βλέπουμε υποχώρηση στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να μας ανησυχεί, διότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο με τον οποίο έχει οικοδομηθεί και θα πρέπει να τα ενισχύουμε και όχι να οπισθοχωρούν. Ε, είναι κρίσιμη η κατάσταση στις χώρες ε, που ζούμε. Ε, το λένε αυτό διάφορες οργανώσεις και το τεκμηριώνουν και το αναγνωρίζει πολύ καλά το σχέδιο έκθεσης που σήμερα συζητούμε. Η Πράσινη και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θεωρούμε ότι η έκθεση θα πρέπει ε, να ξεπεράσει ε, το απλό κατάλογο, την παράθεση που τα γνωρίζουμε αυτά τα δικαιώματα. Θα πρέπει να αναφέρεται και στις παραβιάσεις και πολλές φορές λόγω δράσης ή αδράνειας κάποιων θεσμών. Και πιστεύουμε εμείς οι πράσινοι ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την ποινικοποίηση των ΜΚΟ στην Μεσόγειο, με την καταστολή που υποφέρουν ε, κάποιες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και στη δράση τους, η έλλειψη προστασίας των δημοσιογράφων και των μαρτύρων ε, δημοσίου συμφέροντος, οι γυναικοκτονίες επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το είπανε και άλλοι και ο Άδης και η κατάσταση των μεταναστών και εκείνων που ζητούν άσυλο. Επίσης, όταν δεν έχουμε διάκριση των εξουσιών, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα ή όταν έχουμε ε, διακρίσεις και ε, μυσαλλοδοξία. Τα τελευταία χρόνια τα διαπιστώνουμε όλα αυτά. Περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεστε ε, στους δρόμους μας. Ε, στις διαδηλώσεις δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Αυτά. Δεν θέλω να επεκτάθω πολύ. Ε, θα πρέπει η έκθεση ε, πραγματικά να αντανακλά όλο το φάσμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για να περιγράψουμε τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να το σκεφτούμε και τελικά να δράσουμε. Αλλιώ δεν έχει κανένα νόημα η δική μας εδώ κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ κυρία Ρίμπα. Από την ομάδα ECR, η κυρία Βυσνιεύσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πλήρης και πολλές φορές κινείται και εκτός θέματος. Δεν είναι αντικειμενική η έκθεση αυτή. Θα πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα του χάρτη. Αλλά αυτό αφορά κρατικές αρμοδιότητες σε σχέση με το δικαίωμα στην άμβλωση και την αναπαραγωγική υγεία. Γιατί είναι θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παραβιάζεται το δικαίωμα στην άμβλωση, γιατί δεν προβλέπεται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο άρθρο 2 ο χάρτης αναφέρει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα στη ζωή και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όρισε, όρισε το εξής, ότι στη σύμβαση από τη σύμβαση κανένα άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί μέσα στα πλαίσια του δικαιώματος στην άμβλωση. Ακόμα και το θέμα στην σεξουαλική εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα δεν μπορεί να γίνει λόγος για παραβίαση ενός τέτοιου δικαιώματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται την αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι κυβερνήσεις και τα κράτη έχουν καθήκον και δικαίωμα να οργανώσουν τα εκπαιδευτικά του συστήματα όπως επιθυμούν. Αυτό αφορά και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν θα έπρεπε να γίνει μνήα σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία στα πλαίσια των παραβιάσεων. Εδώ αναφέρεστε και στο ψήφισμα στις, το, της 14ης Νοεμβρίου 19 ως προς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία. Σας εξηγήσαμε ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην Πολωνία και δεν είναι μια κατάσταση που αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια διάκριση ως προς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Πολωνία. Ως προς το δικαίωμα ασύλου δεν λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη κατάσταση και το πλαίσιο ως προς τις μεταναστευτικές ροές. Θα πρέπει να θυμηθούμε και την εξωτερική διάσταση, γιατί μόνο η πραγματική συνεργασία με τις τρίτες χώρες θα μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και την διακίνηση προσώπων. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε μία από τις προγενέστερες παρεμβάσεις για τον εξτρεμισμό της άκρας ε, δεξιάς. Η Επίτροπος Γιουρόβα είπε ότι ο εξτρεμισμός από όπου και να προέρχεται, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, αποτελεί ένα από τα δεινά της κοινωνίας. Και εγώ είμαι αυτής της γνώμης και δεν θα ήθελα να στιγματίζουμε τους ανθρώπους της δεξιάς που δηλαδή έχουν εντάσσονται στο χώρο της δεξιάς. Δεν μπορώ να δεχτώ μια τέτοια συμπεριφορά. Θεωρώ ότι είναι μια συμπεριφορά εξτρεμισμού. Και άλλα μέλη θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την συζήτηση. Βλέπω θα δώσω το λόγο ε, σε αυτούς που έδειξαν ενδιαφέρον. Ο κύριος Θαρταλέχος. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που κάνατε για αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, που μας παρουσιάσατε. Και κατανοώ πως είναι δύσκολο να γίνει αυτό και να αποφασίσει κανείς τι θα συμπεριλάβει και τι θα αφήσει εκτός. Συγκεκριμένα λοιπόν για το λόγο αυτό με εκπλήσει το ότι αναφέρονται τουλάχιστον τρεις φορές στην Ισπανία. Ανεξάρτητα με τα συμπεράσματα ε, τα οποία μας προτείνεται και για τις οποίες θα καταθέσουμε τροπολογίες όπου χρειάζεται, πιστεύω πως η αντικειμενική βάση της ε, ε, έκθεσης θα πρέπει να είναι η ορθή. Μιλάμε λοιπόν για αυξημένο αριθμό πολιτικών ε, κρατούμενων στην Ισπανία γιατί εκφράζουν τις απόψεις τους στα πλαίσια της ε, θητεία τους. Αυτό είναι απερίφραστα ε, λανθασμένο. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή που να είναι στη φυλακή στην Ισπανία επειδή εκφράζει τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Και αυτή είναι μια κατηγορία η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο είδους έγγραφο θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί αυτό και να είχατε προχωρήσει με συνένεση. Αυτό που είχαμε ήταν αδικήματα τα, στα οποία υπέπεσαν πολιτικοί κατά της ένομης και συνταγματικής τάξης, η οποία αποτελεί και τη βάση προστασίας των δικαιωμάτων μας στο Σύνταγμα. Και κατά δεύτερον, αναφέρεστε ε, στα σύνορα της, περιοχής, της πόλης Σέουτα και Μελίγια, στα σύνορα με το Μαρόκο, και μιλάτε για τις επαναπροωθήσεις που γίνονται εν θερμό ανεξάρτητα με την νόμιμη ανησυχία σας, γιατί κάποιες αρχές μπορεί να εκφράσουν ανησυχίες για την κατάσταση στα σύνορα εκεί, το γεγονός είναι πως μια εβδομάδα, πριν από μια εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσίευσε μία απόφαση για ένα θέμα που είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα που ήταν τα summary returns ή ενθερμό επιστροφές στην Σέουτα και στη Μελίγια και ξεκαθάρισε στην απόφαση αυτή το δικαστήριο πως αυτές οι επιστροφές και οι περιστάσεις υπό τις οποίες έγιναν συμφωνούν απόλυτα και συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν αποτελούν καμία καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτά τα δύο σημεία ως προτεραιότητα και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Η κυρία Πούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ από την Πολωνία είμαι βουλευτής, όπου δυστυχώς ε, έχουμε σε πολλούς τομείς ε, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι γυναίκε δεν ε, προστατεύονται από την ενδοοικογενειακή βία, δεν μπορούν να κάνουν νόμιμα άμβλωση. Για να μην μιλήσω για του αναπήρους, για τους Ρωμά, για τι αγρότησε, για του ηλικιωμένου. Εγώ ε, κατάγομαι από μια περιοχή ε, όπου ε, χαρακτηρίζεται ελεύθερη ΛΟΑΤΚΙ. Το 30% του πληθυσμού ζει σε τέτοιες περιοχές στη χώρα μας ε, ε, ξέρει ο κόσμος στο πετσί του τι σημαίνει μίσος. Είμαι από την Πολωνία και ο συνήγορος του παιδιού λέει ότι... Ο συνήγορος του παιδιού λέει ότι μπορείτε να δέρνετε τα παιδιά σας, επιτρέπετε. Και όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες ε, καταστρέφουν τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα γράψει η έκθεση και να ακρούσει τον κόδωνα κινδύνου για όλους μας. Κυρία Νετβέλτ, μιλήσατε εξ ονόματο κυρίας Παγάσα Ορτοντούα, δεν θέλετε να πείτε και δικά σας λόγια, είπα και δικά μου. Ήθελα απλώ να αποκλειθώ στα όσα είπε η κυρία Φωτίγκα για το ότι δαιμονοποιούνται τα κόμματα της δεξιάς. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όλοι έχουν την ελευθερία της επίθεσής τους. Αλλά θα απαντήσω αν ακούσω ακόμα και κάποιον από τη δική σας ομάδα και το κόμμα σας να λέει εδώ πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και βιασμού. Ναι, θα διαμαρτυρηθώ, γιατί είναι ένα φρίκτο αποτρόπιο ψέμα και με τον τρόπο αυτό παρακινούμε στο μίσος. Δεν είναι ε, θέμα θρησκείας ο βιασμός. Είναι ένα καθολικό πρόβλημα και θα έπρεπε να το αναγνωρίζετε και όχι να το χρησιμοποιείτε για να στιγματίσετε μια ολόκληρη ομάδα του πληθυσμού λόγω ρατσιστικών ε, πεπιθήσεων. Και δεν με ενδιαφέρει αν το κάνω από αριστερά ή δεξιά. Εγώ πάντα θα διαμερτύρομαι όταν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Well, well, well, well. Καλώς, καλώς, οκ. Okay. Αν λοιπόν θέλετε να σχολιάσετε βεβαίως. Έχετε το δικαίωμα, αλλά νομίζω ότι θα ξανανοίξει μια συζήτηση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορείτε να μην προσδίδετε ε, ε, προθέσεις που δεν έχω και δράσεις στις οποίες δεν έχω προβεί. Ανεξάρτητα από το ποια κοινωνία ε, εξετάζουμε, η βία πάντα αποτελεί ένα κακό και θα πρέπει να δακτυλοδεικτούμε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για εγκλήματα που αποδίδονται παρά σε ολόκληρη την κοινωνία, αλλά όχι στη δεξιά. Κυρία Κέμπερ, θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί φαίνεται ότι εδώ είμαστε ε, μαζί έξι χρόνια, αλλά είμαστε ένα σχετικά νέο μέλος στην Ευρώπη τα μέλη της παλαιάς Ευρώπης, ας την πούμε έτσι, της γυραιάς Ευρώπης, δεν θα πρέπει να ε, λαμβάνουν, να αναλαμβάνουν το ρόλο των μεντόρων απέναντι στις ε, χώρες μας. Αν θέλετε κάποια στιγμή μπορούμε να πιούμε έναν καφέ μαζί, αλλά δεν δεχόμαστε να είσαστε οι μέντορές μας. Υπάρχουν ε, δύο αξιολογικές ε, διαφορές μεταξύ του σημείου 5 και 7. Αυτές οι αντιφάσεις θα πρέπει να αποσυρθούν. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο, αλλά πιστεύουμε στην εισηγήτρια. Εάν κάποιος είναι κατά της στηρότητας, της στήρωσης, με συγχωρείτε, και εγώ είμαι κατά της στήρωσης και ή ε, τάσομαι κατά της άμβλωσης και υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν μπορείτε να μου αφαιρέσετε αυτό το δικαίωμα. Στην έκθεση αυτή δεν αναφέρεται η προστασία των χριστιανών στην Ευρώπη γιατί χρειάζονται αυτή την προστασία. Χτες η Επίτροπος Γιούροβα δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Πέρσι ε, έγιναν επιθέσεις κατά χριστιανών. Και αυτό πέντε φορές την ημέρα, πέντε επιθέσεις την ημέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, εάν μιλάμε για βία και για δικαιώματα υπέρ των γυναικών, των Ρωμά, σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους χριστιανούς, οι οποίοι ε, την χάνουν διάκριση όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κυρία Κέμπα, ευχαριστώ. Ε, δεν βλέπω άλλα μέλη να θέλουν το λόγο. Οπότε επιστρέφουμε στην εισηγήτρια για να απαντήσει. Α, όχι. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείτε. Παρακαλώ. Η κυρία Μπάρμπαρα Νόλαν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Θέλετε να μας πείτε την απόψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νάταλι Στόκβελ λέγομαι, συνεργάζομαι με την Μπάρμπαρα Νόλαν ε, στη ε, τμήμα τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα ήθελα να Συγχαρώ την ισχύτρια την κυρία Ντέιλι. Είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση, πολύ ωραία διαρθρωμένη. Εστιάζει σε κάποια κομβικά ζητήματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το έργο. Επίσης ευχαριστώ τους κοιόδης ηγητές και τα μέλη, τα υπόλοιπα ε, για τα σχόλιά του. Εύκολο δεν θα είναι για την εισηγήτρια να συγκεντρώσει ε, όλα αυτά τα στοιχεία. Περιμένουμε την τελική μορφή της έκθεσης. Όπως είπε η κυρία Ντέιλι, Θα μας βοηθήσουν οι εργασίες σας για τη νέα στρατηγική, για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω στον Οκτώβριο προτιθέμεθα να σας καταθέσουμε αυτήν τη στρατηγική. Η έκθεσή σας είναι πάρα πολύ σχετική και πάρα πολύ επίκαιρη και εύστοχη. Θα πρέπει να δούμε πώς τα θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω ε, την ε, αλυσίδα των αρχών που καλούνται να εφαρμόσουν ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς αυτής της αλυσίδας, τι εννοούμε, ε, δικαστές, νομοθέτες, διοίκηση, δικηγόρους, κοινωνία των πολιτών, ε, υπερασπιστές, αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, συνήγοροι, διαμεσολαβητές, όλη αυτή η κρίκη της αλυσίδας είναι θεμελιώδης έτσι ώστε να μην παραμένει ο χάρτης κενό γράμμα ή προσδοκίες, ε, όπως είπε η κυρία ε, ε, Ντέιλι, τόσο εύγλωτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπω σα είπα, αν δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο, να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Για να πούμε και το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ, κυρία Ντέιλι. Θα πρέπει καταρχήν να πω ότι δεν θα είναι σύντομη αυτή η συζήτηση όπως πιστεύαμε. Νόμιζα ότι η συζήτηση ήταν πολύ θετική. Χαίρομαι γιατί είχε την επιθυμητή ανταπόκριση. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η εκθέσεις δεν έχουν ε, άμεσο συσχετισμό με μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλη σημασία να δείξουμε τον πολυσχηδή χαρακτήρα αυτής της συζήτησης, γιατί πολλές φορές μιλάμε υπογενικούς όρους. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Βεβαίως υπάρχουν ε, πολιτικές διαφορές αλλά και γνώμες δεν θα ήθελα να μιλήσω ως προς τις πολιτικές ε, διχογνωμίες. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να έχουν τη γνώμη τους, να αντιτάσσονται, αλλά δεν μπορείτε να επιβάλλετε αυτή την άποψη σε άλλους. Και αυτό ε, αφορά και την αντίφαση που είπατε όταν ε, μιλήσαμε για στήρωση αφενός σε ένα σημείο και το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση. Όμως αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα μπορεί να ελέγχει το σώμα της, άρα θα αποφασίσει πότε θα έχει παιδιά και πότε δεν θα έχει. Αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το έχει τονίσει αυτό ιδιαίτερα ως προς την ε, παραβίαση δηλαδή των ε, δικαιωμάτων των γυναικών. Όλα αυτά βασίζονται σε γεγονότα και αυτά προσπαθήσαμε να τονίσουμε. Δεν θα απαντήσω σε σημεία λεπτομεριών, θα το δούμε αυτό συλλογικά και θα λάβουμε υπόψη τα πραγματικά στοιχεία. Θα πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι όταν ε, κατονομάζουμε χώρες, αυτό είναι σίγουρο και χαίρομαι γιατί υπήρξε γενική συμφωνία ως προς την ε, σημασία των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ως προς άλλους τομείς, ως προς τα ψηφιακά δικαιώματα. Θεωρώ, ε, και το έθιξα και στους κοιόδης, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε χώρο σε άλλα ζητήματα. Αν θέλετε όμως μπορώ, μπορώ να ξαναθέσω αυτό το σημείο και εγώ ίδια θα υποβάλω αρκετές τροπολογίες, αλλά όταν κανείς καταρτίζει μία έκθεση θέτει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που μας πλαισιώνει και θα συνεργαστούμε πολύ καλά. Ας δούμε και τις προθεσμίες που έχουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ για αυτά τα καταληκτικά σχόλια. Μπορώ λοιπόν να ανακοινώσω το εξής. Έχει ανοίξει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών Μπορείτε να κάνετε τροπολογίες από τώρα. Επίσης έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Uh, uh, Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 25 Φεβρουαρίου στις 5.30 το απόγευμα. Εντάξει, το σημειώσατε έτσι ώστε να εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεσης στην Επιτροπή Ελευθεριών περί τα μέσα Απριλίου, ίσως 15-16 φέτος. Αυτό είναι ακόμα προς επιβεβαίωση για να πάει στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί η έκθεση το Μάιο. Ενιστό τους έτους. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάνει για ε, το πρωί. Ε, ραντεβού στις 2. Με την ακρόασή μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Γεια σας.